Προχωράμε στην ε, δεύτερη αναγνωσή και στην ε, έκθεση Doyle για τον καθορισμό ορίων καταλήπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και δίνω το λόγο στην κυρία Doyle. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω κύριε Πρόεδρε ευχαριστώντας όλους τους ισχυώδεις εισηγητές οι οποίοι διευκόλυσαν λύναν μία συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση. Πρόκειται για μία τεχνική πρόταση σχετικά με το ισχύον καθεστώς στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσει τους κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων μέσω των τροφίμων καθορίζοντα προέλευσης ε, καθορίζοντας ε, επίπεδα ασφαλείας και ανώτατα επίπεδα για κατάλοιπα για ορισμένες δραστικές ουσίες οι οποίες δεν είναι ασφαλείς ή όπου δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε αν ε, προσφέρουν ασφάλεια. Οι καταναλωτές μπορούν να προστατευτούν εάν υπάρχει παρακολούθηση πριν από τη και χρησιμοποιείται ένας υψηλός βαθμός ασφαλείας για να μπορέσει να παρακολουθηθεί η εξέλιξη του προϊόντος. Συμφωνήσαμε ως προς τα βασικά θέματα. Καταρχήν ε, ε, όσον αφορά τις φαρμακολογικά δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται είτε στο ένα είτε στην άλλη περίπτωση. Δεύτερον, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και παρακολούθηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Μπορέσαμε να διευκρινίσουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εάν ε, βρεθούν ε, μη εγκεκριμένε ουσίες είτε σε ευρωπαϊκά τρόφιμα είτε σε εισαγωγές τρίτων χωρών και υπάρχουν σημεία αναφοράς για δράση δηλαδή τα ανώτατα επίπεδα ε, για τις μη εγκεκριμένες ουσίες. Ε, το θέμα του καθορισμού των ε, ουσιών αυτών για διάφορα απολυμαντικά και άλλες ουσίες έχουν καταρτιστεί και ε, ο καθορισμός ε, της ε, φαρμακολογικά δραστικής ουσίας απαιτεί πολλές έρευνες που δεν είναι δυνατές και ανεκτές για πολλά είδη διότι υπάρχουν ελάχιστοι μικροί χρήστες. Βεβαίως ο καθορισμός αυτός πρέπει να είναι το πρώτο στοιχείο προτού υποβληθεί η αίτηση για έγκριση των, ε, της χρήσεως αυτών ε, των ε, θεμάτων. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί γρήγορα διότι διακινδυνεύει την ασφάλεια των τροφίμων. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε πάντοτε να θεραπεύσουμε ένα ασθενές ζώο αλλά χωρίς να χρησιμοποιήσουμε παράνομη ιατρική. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία περίοδος κατά την οποία θα ε, καθορίζεται ο χρόνος αποσύρσεως ενός φαρμάκου και ο οργανισμός φαρμάκων έχει καθορίσει ε, τα κατάλοιπα για διάφορα είδη μετά το 1997 μετά πειραμάτων πενταετίας κατέληξαν ότι δεν χρειάζονται κατάλοιπα επίπεδα για τα κατάλοιπα για ιδιαίτερα είδη διότι θα έπρεπε να ισχύουν ε, ίδια για όλα τα ζώα. Είτε είναι σημαντικά είτε όχι. Υπάρχουν λοιπόν ε, ε, επίπεδα εκτός από τα εγωπρόβατα και τα, τους χείρους αλλά διαφορετικά το 2008 μετά από εμπειρία 8 ετών έχει καταρτιστεί μία νέα οδηγία η οποία περιγράφει την ε, εφαρμογή της ε, χρήσεως μεταξύ διαφόρων ειδών και επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν σε ε, ό,τι ουσίες χρησιμοποιούνται για τρία βασικά είδη σε όλα τα είδη ζώων ε, διότι επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τις επιπτώσεις της ε, κτηνιατρικής και των σχετικών φαρμάκων. Ε, για τα υποειδή ενδιαφέρομαι προσωπικά και επίσης για τις, τα κλινικά ε, ωφέλη αν δηλαδή πρέπει να είναι ουσιώδης ουσία η οποία χρησιμοποιείται για τα υποειδή. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες για τα υποειδή θα πρέπει να υπάρξει μία περίοδος αποσύρσεως 6 μηνών και θα παρακολούσα την, ε, ε, τον πρόεδρο να σημειώσει η Επιτροπή ότι έπρεπε να αναλάβει να κάνει μία αναθεώρηση ε, των κτηνιατρικών φαρμάκων. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές. Η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις ανώτατες τιμές για τα κατάλοιπα φαρμακολογικά δραστικών ουσιών ε, όσον αφορά ζωικής προέλευσης ε, προϊόντα. Είναι σημαντική η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει στους καταναλωτές από τέτοιου είδους κατάλοιπα φαρμάκων να τους προστατέψει με τα τρόφιμα και ταυτόχρονα η δυνατότητα όσον αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα να βελτιωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και ένα σημαντικό στοιχείο στην ε, απλούστευση του νομικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλούστευση των διεργασιών. Το Συμβούλιο και η Ευρωβουλή ήδη πέρυσι μπόρεσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που αυτή την κοινή θέση που στην κοινή θέση βρήκε τον, την απήχησή της. Έχουμε λοιπόν μια κοινή θέση στην οποία έχουμε καταλήξει και του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της προτάσεις τροποποίησης τροπολογίες και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μπόρεσε να τις δεχθεί, διότι και το πνεύμα και την ουσία της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την διαφύλαταν και την βελτίωναν. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωση προς το, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 8 Ιανουαρίου 2009 <clears throat> εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη όσον αφορά την κοινή θέση. Η έγκριση της κοινή θέσης θα είναι πλέον ε, εφικτή και θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση αυτού του χαρτοφυλακίου πριν από την εκπνοή της ε, κοινοβουλευτικής θητείας αυτού του, ε, αυτής της Ευρωβουλής. Αυτή η ολοκλήρωση θα διευκολύνει τη δουλειά εκείνων που, έχουν, ε, που συσχετίζονται καθημερινά με τέτοιου είδους ελέγχους και κτηνιατρικών προϊόντων και τροφίμων για καλύτερη ε, προστασία και των ε, προϊόντων αυτών και των τροφίμων και εκείνοι που καθημερινά ασχολούνται με αυτό ανέμεναν, προσδοκούσαν με ιδιαίτερη ανυπομονησία να υπάρξει τελική ρύθμιση για τα κατάλοιπα. Και νομίζω ότι σε αίσιο πέρας, πέρας κατέληξε αυτή η προσπάθεια και τώρα επιτέλους βρέθηκε αυτή η λύση προς ικανοποίηση όλων. Γνωρίζω την ιδιαίτερη σημασία της διαθεσιμότητας των φαρμάκων στον τομέα της κτηνιατρικής και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρα από την πρόοδο που σημειώνεται με, αυτή την, με αυτόν τον κανονισμό όσον αφορά τις ανότητες ε, τιμές, ε, όσον αφορά φαρμακολογικά προϊόντα, το 2010 θα έχουμε μια αξιολόγηση των προβλημάτων και επανεξέταση αυτής της οδηγίας όσον αφορά τα φάρμακα στον τομέα της ιατρικής και εκεί όπου θα είναι αναγκαίο και ενδεδειγμένο θα υποβληθούν νέες ε, αναθεωρητικές νομικές, νομοθετικές προτάσεις. Ιδιαίτερε ευχαριστίες πρέπει να εκφράσω εδώ προς την εισηγήτρια σε αυτό το σημείο, προ την κυρία Ντόιλ, για την άοκνη προσπάθεια που κατέλαβε, κατέβαλε και με κάθε τρόπο προσπάθησε να επιτευχθεί η συμφωνία σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Και πάλι ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική σας δουλειά κυρία Ντόιλ. Ευχαριστώ. Ε, κανονικά υπάρχει διαδικασία catch the eye. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν με το catch the eye. Δεν παρακολουθούν οι οθόνες οι οποίες και αυτές έχουν κουραστεί. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει διαδικασία catch the eye θέλει ο εισηγητής να προσθέσει κάτι άλλο. Όχι. Κατόπιν αυτού θα ζητήσω από την εισηγήτριά μας ε, να συνοψίσει. Ευχαριστώ. Όντως κύριε Πρόεδρε κοιτάζω τις σημειώσεις μου, απλώς πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μία τροπολογία την οποία δεν στηρίζω γιατί θα δημιουργήσει ένα νομικό αδιέξοδο, διότι αν δεν υπάρχει μία δοκιμή για να καταρτιστούν τα ελάχιστα επίπεδα, τι θα γίνει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τη βοήθειά της σε αυτό τον τομέα διότι ε, θέλω να σας πω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο αυτή για να αναθεωρήσουμε διάφορες δυνατάξεις για την κτηνιατρική ε, διότι ο τομέας αυτός έχει πολύ ε, προβληματικό προβληματίσει ε, την κοινωνία τα τελευταία χρόνια και οι κτηνίατροι χρειάζεται να εξετάσουν την δυνατότητα υπάρξεως καταλήλων φαρμάκων. Παρ' όλα αυτά όμως η κατάσταση επιδεινώνεται και πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των καταναλωτών, την ευμερία των ζώων και ε, εάν τα ζώα δεν ε, θεραπευτούν με το σωστό φάρμακο ενδέχεται οι ζωονόσινες να έχουν επιπτώσεις και για τους κατοίκους και για τα ζώα και για ε, τα κράτη οπότε ε, γενικώ ένα πολύ βασικό σημείο είναι ότι ε, με τις νέες μεθόδους μειώνονται οι ε, ε, ε, απικίες των μελισσών και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις για την ευμερία πολλών ζώων, για την ασφάλεια της διατροφικής αλυσίας και πρέπει να καλύψουμε τους στόχους της Λισαβόνας, να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες ευρωπαϊκής γεωργίας και να προωθήσουμε την φαρμακοβιομηχανία στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ όλους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Κυρία Ντόιλ, κλείνει η συζήτηση και θα γίνει ψηφοφορία αύριο Πέμπτη. Ε, τώρα λοιπόν έχουμε την ε, έκθεση του κυρίου Τάκουλα σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών για τέσσερα λεπτά.